Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Κοιτάξτε, πολλοί από εσά δεν ψηφίζετε παρακαλώ. Είμαστε την τελική ευθεία παρακαλώ να ξεκινήσουμε τον έλεγχο πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, τελική σκέψη Q υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο. Α κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται, ζητώ συγγνώμη. Η τελική σκέψη R του αρχικού κειμένου. Διαντάσει ρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τελική σκέψη S του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τελική σκέψη V διονομαστικής κλίσεως που άρχεται. Πέρας Απορρίπτεται. Ονομαστική κλίση, τελική σκέψη. Χ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται με δύο ψήφους. Πριν τελική ψηφοφορία, συνάδελφοι, Σα παρακαλώ, εκείνοι που δεν θα συμμετάσχετε στις επεξηγήσει ψήφων, αν έχετε την καλοσύνη να αποχωρήσετε από το μικύκλιο, ώστε να προχωρήσουμε τι επεξηγήσει ψήφων ε, με έναν τρόπο ρυθμισμένο το ψήφισμα σύνολό του να ψηφίσουμε διανομαστικής κλίση που άρχεται πέρας το ψήφισμα ενεκρίθη συγχαρητήρια και σε ένα λεπτό θα συνεχίσουμε τι επεξηγήσει των ψήφων παρακαλώ εκείνους που δεν θα συμμετάσχουν παρακαλώ να αποχωρήσετε με ησυχία Colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στι αιτιολογήσει ψήφου. Καταρχά, επί τη εκθέσεω Βάντεν Κάμπ για την αυτόνομη οδήγηση. Ένα λεπτό καταρχά, η κυρία Μάγερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την έκθεση την αυτόνομη οδήγηση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα τη χαρά να επισκεφθώ ο πρόεδρος Διακόπτη Παρακαλώ, κύριε Μάγερ, λέει ο πρόεδρος. Θα σας ξαναδώσω το λόγο και μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή. Παρακαλώ όμω τους συναδέλφους για μια ακόμη φορά να αποχωρήσουν ησύχω διότι να δίνουν τον ακουστή ομιλήτρια. Κυρία Μάγερ, έχετε ένα λεπτό, μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Χαιρετίζω αυτή την έκθεση για την ε, αυτόνομη οδήγηση. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα πήγα στο Bedfordshire, στο Millbrook, στη δική μου περιφέρεια, που έχει επενδύσει στην υποδομή για την ε, προώθηση των υποδομών για την αυτόνομη οδήγηση. Ένα τεχνολογικό μέλλον ε, μας περιμένει όπου θα είμαστε εμείς χαλαροί και θα μας μεταφέρουν τα οχήματα με ασφάλεια στον προορισμό μας χωρίς ε, τροχέα, χωρίς ε, συμφορήσεις κυκλοφοριακές. Βέβαια θα πρέπει και η επικοινωνία να βελτιωθεί και όλα τα οχήματα θα πρέπει να μιλούν την ίδια γλώσσα. Δεν θα υπάρχουν καμπίνες διερμηνίας ή ακουστικά, επομένως εάν δεν μπορεί να συμφωνήσει η βιομηχανία τα δικά της πρότυπα, θα πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρετίζω ιδίω την πρόταση η Κομισιόν να προτείνει ένα αριθμιστικό πλαίσιο ε, για την V2X συνδεσιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Μέσερ Σμιτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σαν όχημα χωρί οδηγό εδώ και καιρό. Χάρη ε, στην Αμερικανική βιομηχανία και τις ε, εξελίξεις θα έχουμε κάτι που θα διευκολύνει τη ζωή μας ε, στην Ευρώπη. Αυτό βέβαια απαιτεί ρυθμίσεις και κανονισμούς και από ευρωπαϊκής πλευράς δεν γνωρίζουμε ακριβώς ούτε ποιο θα θα είναι το ελισμικό, ούτε το λογισμικό Κάπως αβασάνιστα έχουμε συμφωνήσει να προχωρήσουμε. Θα διαβάζω την εφημερίδα μου και θα με μεταφέρει ένα αυτοματοποιημένο όχημα στο μέλλον. Να δούμε όμως τι γίνεται και με τι εμπειρίες από τη σύπα με κάποια ατυχήματα και με τα πειράματα που έχουν γίνει και... Ο κύριος Τρογεύσκη για ένα λεπτό είναι ο επόμενος ομιλητής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη συζήτηση που κάναμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αυτόνομα εξοπλιστικά συστήματα. Τώρα έχουμε την αυτόνομη οδήγηση, αλλά αποφεύγουμε αποτελεσματικά το νομικό ζήτημα. Ε, την έκθεση και το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει, προβληματίζομαι. Ε, πιστεύω ότι και αυτή τη φορά δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο. Για την έκθεση δεν είχαμε μεγάλες διαφορές. Έγινε με μεγάλη πλειοψηφία δεκτή έκθεση και ελπίζουμε ε, μέχρι το 2022 να έχουμε ετοιμάσει τις νομικές διατάξεις που θα μας ε, ε, διασφαλίζουν απέναντι στις αρνητικές συνέπειες της τεχνολογικής εξέλιξης. Για ένα λεπτό τώρα, το λόγο κύριος Χάουαρθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω την έκθεση και την προσέγγιση της Επιτρόπου Γιούροβα που μας την παρουσίασε χθε το βράδυ. Τρεις πυλώνες ε, γύρω από το νομικό πλαίσιο χρηματοοικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη των τεχνολογιών, κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις ε, της αυτόνομης οδήγησης. Ε, υπάρχουν τα αισθήματα της αστικής ευθύνης και η ανάγκη να προσαρμοστεί η τεχνολογία. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν. Υπάρχει επιθυμία σαφής ε, από τεχνολογικές εταιρείες όπως ε, Amazon, Google να ε, δαπανίσουν πολλά κονδύλια. Αλλά υπάρχει ένας τέταρτος πυλώνας που είναι η δημόσια αποδοχή των αυτόνομων οχημάτων. Είναι ε, σημαντικό όμως ε, να δοθεί στην ασφάλεια. Έχουμε ίσως τον αυτόματο πιλότο στις, αυτομετα... στις ε, νέες μεταφορές, όμως τα, τα οχήματα είναι κάπως πιο προσωπικό ζήτημα. το θέμα είναι λοιπόν να διαρωτηθούμε, θα μπορώ στο μέλλον να οδηγήσω το δικό μου αυτοκίνητο ή όχι. ο μιλητής. Ο κύριος Σέινφελτ, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, παρατηρούμε ε, τελευταία πολύ δυναμική ανάπτυξη του ψηφιακού τομέα. Και είναι μία αναστρέψιμη αυτή η διαδικασία. Λαμβάνοντα λοιπόν υπόψη τι ραγδαίε τεχνολογικέ εξελίξει, θα πρέπει και η Ευρώπη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Για να συμβεί όμω κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνουν και απαραίτητε επενδύσει, κυρίω στι υποδομέ, στι οδικέ μεταφορέ, αλλά και στην ηλεκτρονική διασύνδεση των ευρωπαϊκών ε, οδών. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και την απαραίτητη κανονιστική νομοθετική ρύθμιση και την, ε, ε, τον επιμερισμό των ευθυνών σε περίπτωση ε, αυτοματοποιημένη οδήγηση. Τι θα γίνει σε περίπτωση που τρακάρουν τέτοια αυτοματοποιημένα οχήματα. Θα πρέπει να, αξιολογήσουμε, να αξιοποιήσουμε την, τεχνική την νομοποίηση αλλά με την κατάλληλη νομοθετική οριοθέτηση. Και φυσικά θα πρέπει να αποφύγουμε και αρνητικά κοινωνικά αποτελέσματα σε τέτοια ανάπτυξη μαζικής ε, προσέγγισης. Κυρία Κλούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόσδεκτη αυτή η έκθεση. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό που αφορά την ανάπτυξη του συστήματος και τι ωφέλη μας δίνουν τα αυτόνομα οχήματα, τα οχήματα χωρίς οδηγό. Θα μπουν στην αγορά μετά το 2020 και γρήγορα μάλιστα. Και μετά θα επεκταθούν και σε φορτηγά και διάφορα άλλα μεγάλα οχήματα, αν πάνε καλά τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά θέματα προ εξέταση, αν θέλουμε να έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές. Θέλουμε να δούμε την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των στοιχείων. Και βέβαια την ασφάλεια των ανθρώπων. Τεχνικά πρότυπα χρειάζονται για τα οχήματα και τι υποδομέ. Χρειάζεται να, έχουμε, να εξετάσουμε ποιο είναι υπεύθυνο, ποια είναι τα δεντρολογικά θέματα Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε στον τομέα, υπάρχουν πολλά ερωτήματα προς απάντηση και μπορούν να γίνουν εδώ και στα Εθνικά Κοινοβούλια και να γίνει ε, αποδεκτή αυτή η έννοια των αυτονόμων ηχημάτων από όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ο κ. Πολτσακ. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η έκθεση είναι πολύ σημαντική ε, το θέμα είναι ευρύτατο. Υπερψήφισε την έκθεση, ενδιαφέρει την αυτοκινητοβιομηχανία, την ψηφιακή οικονομία, την καινοτομία και αναφέρεται και στο ζήτημα της μείωσης των καυσαερίων. Είναι αναφιβολό ότι θα πρέπει να δώσουμε ναύσματα και κίνητρες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να στηρίξουν αυτό το κλάδο ώστε να γίνουμε φορέα καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να φτάσουμε και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού με τις δικές μας τεχνολογίες και καινοτομίες. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία του κλάδου, ε, ιδιαίτερα στα θέματα της αυτόνομης οδήγησης και των αυτοματοποιημένων οχημάτων. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και το ζήτημα της ε, συνδεσιμότητας ε, των συνδεδεμένων οχημάτων. Θα πρέπει φυσικά για τα θέματα αυτά να ασχοληθούν και οι περιφέρειες στα πλαίσια και των τοπικών μεταφορών. Ο κύριος Χάναν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Την επόμενη φορά θα είστε σε μια πόλη, ρίξτε μια ματιά γύρω σα. Μετρήστε. Πόσοι οδηγούν για να ζήσουν. Οι οδηγοί λεωφορείων, των φορτηγών, των Uber, των ταξί. Αφήστε του και θα δείτε ότι είναι ο μεγαλύτερο συλλογικό εργοδότης τα αυτοκίνητα. Όταν γίνουν τα αυτόνομα αυτοκίνητα αυτό, ε, πραγματικότητα θα χαθούν πολλέ δουλειέ σε αυτό το τομέα. Και αυτό οδηγεί σε κάποιε ανησυχίε που ακούστηκαν στο Κοινοβούλιο δεν συνεπάγεται ότι όλοι αυτοί θα τριγυρνάνε άνεργοι αυτοί οι άνθρωποι. Εάν δούμε σήμερα που είναι όλοι άνεργοι ε, αυτοί που δούλευαν στα βίντεο κλαμπ, οι γραμματείς, οι αρχιοθέτες. Η τεχνολογία ένα αλλάζει και όμως περισσότεροι άνθρωποι ε, δουλεύουν στις χώρες μας τώρα, περισσότερο τώρα παραποτέ στην ιστορία. Ίσως η τεχνητή ευφυΐα και οι σύγχρονε τεχνολογικέ αλλαγέ οδηγούν σε αυτό. Αυξάνεται το επίπεδο διαβίωση και δημιουργούμε νέε θέσει απασχόληση, ενώ οι συνθήκε βελτιώνονται. Ρίξτε μια ματιά γύρω σα και κοιτάξτε πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε αυτή την εποχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ, κύριο Σκέλη τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση διότι πιστεύω πως είναι ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο η αυτόνομη οδήγηση, γιατί απαιτείται δουλειά, απαιτείται πρόοδο. Πρέπει να γίνει για να φτάσουμε χώρε όπω είναι η ΕΠΑ, η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, που προπορεύονται οι μόνε ό,τι αφορά και την έρευνα και τι ρυθμίσει. Η αυτόνομη τεχνολογία στον τομέα των μεταφορών και τη ευαδιαστική αλυσίδα είναι σημαντικό, προσφέρει σημαντικό δυναμικό ε, για το μέλλον, για το οδικό δίκτυο Μπορεί να βοηθήσει αυτό και την οικονομία και την κοινωνική ζωή. Η χρήση drones για τη μεταφορά αγαθών, ε, τα ευφύ συστήματα σηματοδότηση για τη συγκοινωνία στις πόλεις ε, και τα οχήματα με λειτουργικέ δυνατότητες αυτόνομη οδήγηση ε, είναι στη γωνία, είναι στο άμεσο μέλλον και ελπίζουμε να γίνουν πραγματικότητα και να χρηματοδοτηθούν ιδίω στο πλαίσιο του επόμενου ορίζοντα προγράμματος αυτού πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Πρόεδρος, να προχωρήσουμε στην επόμενη έκθεση για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Μέσερ Σμιτ για ένα λεπτό πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Στις εκλογές ε, του 2014 οι οδικές μεταφορές και οι μεταφορές εν γέννη ήταν ένα από τα σημαντικά ζητήματα. Ε, το καμποτάζ ήταν μια, γλώσσα, μια λέξη που οι Δανείοι την χρησιμοποίησαν καθημερινά ε, και στην προεκλογική συζήτηση. Πώς μπορεί κανείς να είναι σε μια χώρα μέλος αλλά να εργάζεται σε μια άλλη χώρα μέλος. Αθέμπτος ε, ανταγωνισμός που μπορεί να προκύψει Ωστόσο υπήρχαν και προσδοκίες για το καμποτάζ. Υπήρξε κόσμος ο οποίος απογοητεύτηκε όταν είδε ότι δεν έγινε τίποτα. Ή αν κάτι έγινε αυτό ήταν στη λάθος κατεύθυνση. Άρα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν είναι στην τροχιά που θα έπρεπε. Πόρο απέχουμε της πραγματικότητας. Στις 28 Οκτωβρίου του 2018, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών μας ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο δεν θα είναι έτοιμο για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την έκθεση αυτή. Η έκθεση αυτή τελικά έγινε δεκτή ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Αρμόδια Επιτροπή και μάλιστα οι τροπολογίες 28 και 34 δυστυχώς καταστρέφουν, αλλοιώνουν αυτή την έκθεση. Οι υπόλοιπες τροπολογίες και οι αρνητικές ε, τελικά απορρίφθηκαν. Γι' αυτό έχουμε καλό σημείο αφετηρίες. Ε, περιμένουμε όμως την απόφαση στο Συμβούλιο. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ασκήσουμε πιέσεις ε, όσο γίνεται, ώστε να γίνει osonoύπο δεκτή η πρόταση, γιατί πρόκειται για πολύ σημαντική δραστηριότητα ενός πολύ σημαντικού κλάδου της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Σέινφελτ. Ευχαριστώ. Εδώ και δεκαετίες προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την ενιαία αγορά στην Ενωμένη Ευρώπη. Δυστυχώς όμως, παρά το πέρασμα πολλών ετών, η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και η ελεύθερη διακίνηση προσώπων ε, ε, έχει πολλέ ρυθμίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλέ ρυθμίσει που περιορίζουν την ελεύθερο ανταγωνισμό, την οικονομία, την ελεύθερη διακίνηση και κυκλοφορία και παρεμποδίζουν και την ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι υπερβολικέ κανονιστικέ ρυθμίσει. Εγώ είμαι υπέρμαχο τη φιλελευθερωποίηση ε, για τη χρησιμοποίηση ε, των ε, μισθωμένων οχημάτων χωρί οδηγό. Πιστεύω ότι η απελευθέρωση τέτοιων διατάξεων θα εξυπηρετήσει όχι μόνο τις μεταφορές, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη, γιατί θα εξασφαλίσει θέσεις απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών. Επίσης, είμαι κατά των περιορισμών που προκύπτουν από το πακέτο της κινητικότητας που εξετάζουμε τον τελευταίο καιρό στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάναν έχει ε, φύγει, οπότε δεν θα χρειαστεί να ακούσουμε τη δική του επεξήγηση ψήφου. Περνάμε στην επόμενη έκθεση. Ο κύριος Μέσσερ Σμιτ για την έκθεση Μλίναρ σε ό,τι αφορά τη συνεκτίμηση τη διάσταση του φίλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συζήτηση για ε, επανειλημμένα ψηφίσματα για την ισότητα των φύλων ή για την συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, αλλά παρόλα αυτά τα πράγματα δεν κινούνται με τη δέουσα ταχύτητα. Στην ε, δεν έχουμε την πρόεδρο της Βουλής γυναίκα, η Πρωθυπουργό είναι γυναίκα, η, μας, η Επίτροπός μας είναι γυναίκα, για να μην μιλήσω για τη Βασίλισσά μας που επίσης είναι γυναίκα. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι η πρόεδροι και των τριών θεσμικών οργάνων και ο πρόεδρος της ΕΚΤ είναι άντρες. Δεν θα πρέπει να τα εξετάσουμε και να τα σχολιάσουμε όλα αυτά στην έκθεση. Δεν θα πρέπει να είναι αυτό το επίκεντρο της έκθεσης. Όχι όμως. Μιλούμε για ε, διατύπωση που θα είναι ουδέτερη από την άποψη του φίλου και μιλούμε για κάποιες άλλες ανοησίες και αντί να πιάσουμε τον, τον τάβρο από τα κέρατα, εμείς μιλάμε και λέμε άλλον. Ο κύριος Πιοτρόφσκι, ευχαριστώ η έκθεση για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σημείο στην παράγραφο 15 μιλά για την αλλαγή της διατύπωσης ώστε να είναι ουδέτερη από την άποψη φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο. Κάτι που δημιουργεί κάποιες, κάποια παράλογα αποτελέσματα που δεν έχουν σχέση με την ισότητα των φύλων. Επίση, ε, παρόμοια δημοσίευση είχαμε το 2008, μάλιστα με τον ίδιο τίτλο. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πολύ γρήγορα αρχιοθετήθηκε το σχετικό ψήφισμα, γιατί κρίθηκε παράλογο σε πολλές χώρες. Επίσης, ε, το σημείο γιου στο προήμιο που μιλάει για τους ΛΟΑΔΜΑ, που δεν έχουν την δέουσα παρουσία. Είμαι φυσικά κατά όλων αυτών των σημείων και γι' αυτό καταψήφισα την έκθεση Μλίναρ. Η κυρία Κρούπα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Και εγώ καταψήφισα την έκθεση Μλίναρ με θέμα την εσωμάτωση της διάστασης φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και καταψήφισα όχι γιατί είμαι κατά της ισότητας των φύλων, αλλά είμαι κατά μερικών ε, παράλογων παραγράφων της έκθεσης. Ιδιαίτερα στην αιτιολογική σκέψη ΑΔ που μιλάει ότι για τη συνεκτίμηση του φύλου θα πρέπει να χρειάζονται ιδιαίτερες ε, δεξιότητες και με θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα διαφορετικά σωματικά ή ψυχολογικά χαρακτηριστικά ή για την ικανότητα, τη βιολογική ικανότητα των ε, γυναικών να γεννούν παιδιά και φυσικά η συμμετοχή τους στην ανατροφή ιδιαίτερα στις πρώτες φάσεις ηλικίας είναι κάτι πολύ απαραίτητο για την ε, υγεία, την ψυχολογική του παιδιού. Και σίγουρα η ισότητα των φίλων είναι θέμα ανθρώπινων δικαιωμάτων, ε, δημοκρατικότητας και κράτους δικαίου. Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα, το τα δικαιώματά τους, να γίνουν μητέρες και να επιλέγουν να αναθρέψουν μόνες τους τα παιδιά τους. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Βυσνιεύσκα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εγώ επίσης καταψήφισα την έκθεση Μλίναρ γιατί περιλαμβάνει κάποιες ε, ε, παραγράφους που με βρίσκουν καθέτα αντίθετη. Επίσης, αναφέρεται ότι θα πρέπει να μην φυστούμε προσπαθειών προκειμένου να καταπολεμήσουμε την σεξουαλική παρενόχληση. Ε, νομίζω ότι ως προς αυτό δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Όλοι είμαστε κατά τη σεξουαλική παρενόχλησης. Όλοι είμαστε κατά της χρήση βίας. Κρίμα όμως που στην έκθεση αυτή δίνεται όλη η έμφαση σε ιδεολογικά θέματα που αφορούν τη μητρότητα, την πρόθεση των ΛΟΑΔΜ και επίσης προτείνεται η ε, ουδέτερη διατύπωση ε, για το θέμα του φύλου. Επίσης, νομίζω κάποιες αριστερίζουσες παρατάξεις θέλουν να επέμβουν και στα θέματα τα γλωσσικά. Αυτό είναι απαράδεκτο, αυτή η παρέμβαση είναι απαράδεκτη. Οι γυναίκες είναι έξυπνες, χρειάζονται ρυθμίσεις που θα τους επιτρέπουν να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ κύριο Σκρίπεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ το νόημα των, το νόημα των λέξεων ισότητα των φίλων έχει αλλάξει από όταν χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξεκινήσαμε με τι διαφορέ των αμοιβών. Μιλήσαμε για διαφορέ στι αμοιβέ όσον αφορά άντρε και γυναίκε που εργάζονται στην ίδια θέση. Είναι μια ισότητα που θα πρέπει να επιληθεί. Μάλιστα, από την άλλη πλευρά, ε, θα πρέπει να εκτιμήσουμε την προσέγγιση των γυναικών στην εργασία. Μπορούν να σκέφτονται διαφορετικά. Ε, μπορούν να συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο. Φέρνουν μια ειρήνη στην εργασία, στι επιχειρήσει και στην πολιτική, όμω δυστυχώ είναι οι πιο επιθετικέ είναι πιο ορατοί οι πιο επιθετικοί. Γι' αυτό φαίνονται περισσότερο οι άντρε, γιατί δεν φοβούνται το να είναι ορατοί οι άντρε. Θα ήθελα να έχουν περισσότερο χώρο για τις γυναίκες εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να ισχυροποιηθούν στο Ευρωκοινοβούλιο γυναίκε. Αλλά μετακινηθήκαμε κάπου στη συζήτηση και τώρα παρακολουθούμε την εκπροσώπηση των γυναικών στου διάφορου φορεί τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δεν μπορούμε να διατάξουμε κάτι. Θα πρέπει να εργάζονται εδώ, αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την χρήση των γυναικών σε αυτά τα όργανα. Πρέπει να τι σεβόμαστε, αλλά θα πρέπει να μιλάμε περισσότερο για τη συμφιλίωση τη οικογενειακή και εργασιακή ζωή. Ο κ. Χάναν δεν είναι εδώ. Ο τελευταίο αγορητή θα είναι ο κ. Κέλλη, όσον αφορά αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε υπερψήφισα αυτή την έκθεση και υποστηρίζω τα διάφορα μηνύματα που αναφέρονται και το γενικότερο μήνυμα που διαβιβάζεται ότι η διάκριση ουδήποτε είδου είναι κάτι απαράδεκτο στο Ευρωκοινοβούλιο. Η ισότητα των φύλων δεν υπάρχει εντό του δικού μα θεσμικού οργάνου και πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ισότητα των φύλων στη γενικότερη, στην ευρύτερη κοινωνία. Καλωσορίζω τα επιτέχματα που επιτέχθησαν τα τελευταία δύο χρόνια, όπω περιγράφτηκαν στην έκθεση. Και πριν τι ευρωεκλογέ, είναι ο κατάλληλο χρόνο να δούμε πού μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσει για την επόμενη θητεία. Ε, μια από τι πιο αξιοσημείωτε δράσει του Κοινοβουλίου που ανελήφθη πρόσφατα ήταν να έχουμε πρόγραμμα κατάρτιση που αφορά του ευρωβουλευτέ πάνω σε αυτά τα θέματα. Εγώ πέρασα, έκανα αυτή την εκπαίδευση και θεώρησα ότι άξιζε τον κόπο. Νομίζω ότι αυτή η εκπαίδευση είναι σημαντικότατη και θα καλούσα όλου του συναδέλφου να συμμετάσχουν. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ισότητα των φίλων. είναι στην πρώτη γραμμή πάντα σε ό,τι κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Οπότε φτάσαμε στην έκθεση Brian Hayes η αξιολόγηση της χρήσης του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα. Η κυρία Σδριεύσκη είναι η πρώτη. Για ένα λεπτό. Ο κύριο συγγνώμη. Ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι αναφυσβήτα σημαντικό εργαλείο του δημόσιου τομέα. Δεν θα ήθελα η επιρροή ε, του κοινοτικού προπολογισμού να αυξηθεί ιδιαίτερω. Και ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι αλλαγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν ισχύει. Το 2007, στην έκθεση που περιέγραφε τα πιθανά αποτελέσματα της μεταρρύθμισης ε, ε, της ε, οικονομικής πολιτικής στα κράτη-μέλη. Δυστυχώς ήταν πολύ επικριτικά τα αποτελέσματα του κοινοτικού προϋπολογισμού και της επιρροής του. Και, και πάλι είδαμε το θέμα της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, της δημόσιας διοίκησης, που μερικές φορές γίνεται ασυνάρτητα, χωρίς συνοχή και χωρίς επικέντρωση στα ουσιώδη. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και στην τελευταία έκθεση την ανάγκη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων σχεδίων και προγραμμάτων, κάτι που δεν ε, υπάρχει. Και επίση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιρροή τη πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν ισχύει επίση. Η συνάδελφο κυρία Νιριάντα; Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπραν Χέις ε, είναι ο συντάξης έκθεση και μέρος του Φίνα και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραματίσει ένα πιο κεντρικό ρόλο στη δημόσια δίκηση των κρατών μελών. Και αυτό παρά το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει νομική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τι εθνικέ δημόσιε διοικήσει. Υπάρχουν μελέτε που δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποιεί ουσιαστικά ε, την ε, αυτές τις προτάσεις που γίνονται για μεγαλύτερη παρέμβαση για να επιβάλλει, για να ασκήσει επιρροή. Ουσιαστικά πρέπει να δοθούν κίνητρα ε, στις χώρες που ε, προωθούν μεταρρυθμίσεις. 25 δις του προπολογισμού θα χρησιμοποιηθούν γι' αυτό στην προσεχή, στην προσεχή επταετία. Ξέρουμε στην Ιρλανδία ότι θα, πρέπει, ε, θα, γίνουν δεκτές αυτές οι αποφάσεις. Υποτίθεται ότι οι κοινωνικές προκές δεν πρέπει να ε, θυγούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, αν πάρει περισσότερη εξουσία, θα ασκήσει επιτροπές ε, πολιτικές τις οποίες υποστηρίζουν τα μεγάλα κόμματα στην ε, χώρα μου και αυτό δεν το υποστηρίζουμε. Ο κύριος Πόλτσακ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ψήφισε υπέρ. Παρότι γνωρίζω ότι ο ρόλος μας πιο πολύ είναι δημιουργία συνεργασιών και παροχή κινήτρων στα κρατη έχουν αυτά την ευθύνη για τη δημόσια Όμως ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να προστατευτεί. Θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να επικοινωνούν με τις δημόσίε διοικήσεις του ε, με τις ψηφιακές τεχνολογίες και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ω αρρώγο. Θέλουμε να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Τις πληροφορίες που αναζητούν μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών και τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έχουμε ένα εργαλείο της πολιτικής συνοχής που εκεί αποσκοπεί και προσπαθεί επίσης να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της δημοσίας διοίκησης. Είναι σαφής εδώ ε, και η σημασία της δημιουργίας υποδομών και ικανοτήτων. Αυτά μας ενδιαφέρουν περισσότερο και θεωρούμε ότι είναι κάτι απαραίτητο αν θέλουν τα κρατημέλη να έχουν επιτυχή δημόσια διοίκηση. Τώρα περνάμε στι κατευθυντήρε γραμμέ Ευρωπαϊκή Ένωση, εντολή του ειδικού απεσταλμένου Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση τη θρησκευτική ελευθερία και τη ελευθερία των πεπιθήσεων εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο τρόπο και ένα λεπτό. Ε, η έκθεση ΞΥΜΠΑ μιλάει για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία πεποίθησης ως ε, αναφέρεται το ανθρώπινο δικαίωμα. Και στην παράγραφο 2 εκφράζουμε μεγάλη ανησυχία για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε βίαιη αύξηση της ε, παραβίασης της θρησκευτική ελευθερίας ή δίωξη των πιστών ανά τον κόσμο. Για παράδειγμα, η Άσια Μπίμπη, αναφέρομαι στο σημείο 13, ζεκαπευθύν ε, με έκκληση στις αρχές του Πακιστάν εξασφαλίσει την ε, ασφάλεια της κυρίας Άσια Μπίμπη. Επίση, ό,τι αφορά την προστασία τη θρησκευτική ελευθερία και τη ελευθερία πεπιθήσεω εκτό Ένωση, ε, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την προστασία των χριστιανών. Δυστυχώ, ε, η έννοια χριστιανό δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο τη έκθεση. Κι όμω οι χριστιανοί είναι η ομάδα που κατεξοχήν διώκεται στον κόσμο και γι' αυτό κράτησε στάση αποχής ε, στην έκθεση XIP. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γιούρεκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Η έκθεση αυτή ε, ξεκινάει ε, από το θέμα της, του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας που είναι συνταγματικό ζήτημα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αυτός είναι υπεραπλουστευτισμός, είναι λαϊκιστική θέση και δεν ευσταθεί κιόλα. Και μάλιστα στην Πολωνία έχουμε αυτονομία και ανεξαρτησία των πολιτικών από τις θρησκευτικέ εξουσίες και επίσης υπάρχει η αρχή της συνεργασίας κράτους και εκκλησίας προς το κοινό καλό και το καλό των πολιτών. Θα πρέπει αυτό να το λάβει υπόψη η έκθεση και το σύνθημα του διαχωρισμού ε, να μην γίνει ως πρόσχημα για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, τις διώξεις, όχι μόνο σε κομμουνιστικά καθεστώτα ή σε χώρες ε, όπως το Μεξικό που εφαρμόζουν τέτοιες διώξεις. Είναι σημαντικό στο δίκαιο να είμαστε πολύ ακριβείς στη διατύπωση. Γι' αυτό είμαι κατά οποιασδήποτε ιδεολογικής προσέγγισης που θέλει να αποκλείσει τους χριστιανούς από τον πολιτικό βίο της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όσνιος έχει το λόγο για ένα λεπτό. Όπως ε, αναφέρθηκε, ξεκινά από ένα ε, ανεδαφικό ε, σχόλιο ότι ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας είναι συνταγματική αρχή σε όλο τον κόσμο. Κι όμως ε, στη, στο, στο Βρετανικό Δίκαιο δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει στενή ε, σύνδεση της Αγγλικανικής Εκκλησίας ε, με το κράτος. Επίσης έχουμε και το Βατικανό. Είναι πολύ ανόητο το προήμιο λοιπόν της έκθεσης που μιλάει για τον συνταγματικό διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Επίσης, αν μιλούσαμε για ομάδες που διώκονται, περιλαμβάνονται δικές, ε, γυναίκες, ΛΟΑΔΜΑ, Απ' τη μια μιλούμε για διώξει και αναφέρουμε ονομαστικά γυναίκε, ΛΟΑΔ, ενώ όταν έχουμε διώξει χριστιανών, γιατί δεν αναφέρουμε και τη λέξη χριστιανό μέσα. Οι διώξει κατά των χριστιανών είναι πολύ πιο έντονε απέναντι στι ε, ε, αρνητικέ συμπεριφορέ κατά φεμινιστικών οργανώσεων. Ε, λυπάμαι λοιπόν που έγινε δεκτή αυτή η έκθεση του κυρίου Ξύπ και όσο την προσυπέγραψαν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ξύπεκ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. 70 χρόνια μετά την έγκριση της Οικουμενικής Διακήρυξης δεν έφτασαν ε, ώστε να τα απολαμβάνουν τα δικαιώματα όλοι. Ελευθερία σκέψη, θρησκευτική ελευθερία. Ε, πλήττονται τα δικαιώματα όχι μόνο των χριστιανών αλλά και άλλων μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή. Στηρίζω λοιπόν ε, αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να βοηθήσει αυτό για την πρόθεση της ανεξιθρησκείας. Πολλοί δολοφονούνται στον κόσμο επειδή θέλουν να συνεχίσουν να επιλέγουν ελεύθερα τα πιστεύω τους, αλλά μπορεί και να, πολλέ... Ε, να επιλέξουν να είναι άθινο, να πιστεύουν σε τίποτα. Ασέα Μπίμπι πρέπει να απελευθερωθεί Το προσπαθούσε να ξεφύγει ε, από τα βασανιστήρια στο Πακιστάν και ε, είναι εκεί κάπου στη χώρα. Ε, υπάρχουν ε, πολλοί οποίοι διώκονται για τα πιστεύω τους. Έγινε λόγος και για τον ειδικό απεσταλμένο για την πρόσθεση της κεφτικής Πράγματι πρέπει να ενταχθεί στην εξωτερική μας πολιτική το έργο αυτό του απεσταλμένου. Επόμενο και τελευταίο θέμα, ισότητα των φίλων και πολιτικές. Κυρία Μάγερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχει, γίνει, έχει επικρατήσει μεγαλύτερη ησυχία. Μηδενικό φόρος ε, για τα ε, σερβιέτε και τα ταμπόνα. 18.000 ε, ε, λίρες ε, δαπανά το χρόνο η γυναίκα για την εμεινορίση που συμβαίνει κάθε μήνα και υπάρχει στίγμα της περίοδου στη Ηνωμένο Βασίλειο μία στις 10 γυναίκες δεν μπορούν να αγοράσουν σερβέτες και ταμπών και κάποιες γυναίκες κορίτσια δεν μπορούν να πάνε καν σχολείο λόγω αυτού μιλάω για το στίγμα διότι Πολλέ γυναίκε βιώνουν την εμμενορίση του ε, στα κρυφά ω ταμπού. Καλό τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει ε, να παρέχουν ε, αυτά τα είδη δωρεάν όπως θα πρέπει να γίνεται και με το χαρτί υγείας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιοτρόφσκι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η ομάδα ECR καταψήφισε την έκθεση Ματίας Ουρτασούν γιατί κατά τη γνώμη μας πολύ εσφαλμένα παρουσιάζεται η φορολογική πολιτική των κρατών μελών ως πολιτική που συνιστά διακρίσεις. Στο σημείο 1 αναφέρεται η καταπολέμηση του φαλοκρατικού μοντέλου και της οικογενειακής οργάνωσης και ζητά η κατάργηση οποιαδήποτε φορολογικών δαπάνων που, δαπανών που ε, συνδέονται με τα κοινά έσοδα. Επίσης, ε, το ΕΛΚ ε, άσκησε πολλές επικρίσεις κατά της έκθεσης ε, ενώ δεν ε, γίνεται σεβαστό το δικαίωμα επιλογής του φορολογικού συστήματος ε, και τη προστασία τη οικογένειας. Για όλου αυτού του λόγου καταψήφισα την έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Κρούπα για ένα λεπτό. Και εγώ ψήφισα κατά της έκθεσης με θέμα την ισότητα των φύλων στη φορολογική πολιτική. Παρόλο που είμαι υπέρ του ίσου μισθού για την ίση εργασία, και είμαι υπέρ τη ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και είμαι υπέρ τη καταπολέμησης των διακρίσεων. Δεν θεωρώ όμω ότι θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα επιλογής του φορολογικού συστήματος για τις ευρωπαϊκές οικογένειε. Και η εξατομικευμένη φορολογία, η ξεχωριστή φορολόγηση ε, είναι ουσιαστικά εις βάρος της οικογένειας, ε, καταπολεμάται και παραβιάζεται η επικουρικότητα, η αναλογικότητα και μερικές φορές είναι άδικη μια τέτοια επιβολή για τις γυναίκες γιατί η, σίγουρα η δημιουργία οικογένειας και η ανατροφή των παιδιών είναι στο αγαθό και δικαίωμα των γυναικών ενώ αντιμετωπίσει τις γυναίκες ως εργατικό δυναμικό όταν εργάζονται στην οικογένεια αποτελεί άρνηση του φυσικού και βιολογικού ρόλου της γυναίκας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όσνιες, για ένα λεπτό. Έχουμε άλλη μια έκθεση που χαρακτηρίζεται από την ιδεολειψία του φίλου και χαρακτηρίζει την κοινοβουλευτική πραγματικότητα δυστυχώς. Επίσης, ε, μιλούμε ε, για τα για τη δυνατότητα, για, την, ε, για τη μεγαλύτερη οικονομική ε, άνεση των ανδρών που έχουν και τα περισσότερα κίνητα και τι είναι και τι λόγο ε, έχετε που το αναφέρετε κάτι τέτοιο ακόμη και αν υπάρχει, αν ισχύει, αν ισχύει αυτό. Δεν θέλουν οι γυναίκε να είναι ιδιοκτήτριε ακινήτων μερικέ φορέ. τι θα πρέπει να του αναγκάσουμε να το κάνουν. Τι, τι θα πει αυτή η έκθεση που λέει ότι οι άνδρε περισσότερο είναι ιδιοκτήτε ακινήτων. Συμφωνώ ε, ότι η φορολογία έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Φυσικά δεν ισχύουν τα ίδια πραγματικά περιστατικά, οπότε γιατί να έχουμε τις ίδιες φορολογικές διατάξεις. Ανάλογα με το φύλλο έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις, ε, διαφορετικές, ε, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορείτε με το στανιό να επιβάλλετε μια ισότητα ή εξομοίωση των χαρακτηριστικών. Ευχαριστώ. Η κυρία Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ παρόλο που είμαι υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών, δεν μπόρεσα να υπερψήφισω την έκθεση που θέμα έχει την ισότητα των φύλων στα πλαίσια της φορολογικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η έκθεση περιλαμβάνει εξτρεμιστικές, αριστερίζουσες απόψεις που δεν είναι καθόλου αντικειμενικές. Αναφέρεται ότι η, η διάκριση αυτή είναι γενική και χρειάζεται μια ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση των φορολογικών ε, πολιτικών των κρατών μελών για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Διαφωνώ με αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι μεροληπτική και υποκειμενική αυτή η άποψη. Αντί να μιλούμε για ισότητα ανδρών και γυναικών, παρουσιάζεται ένα όραμα και μια προσέγγιση τη δική σας ε, για τα δύο φύλλα. Αυτή η προσέγγιση σας ε, συνιστά διακριτική μεταρρύθμιση. Γιατί αντί να στηρίζετε τις γυναίκες και να τις δίνετε ευκαιρίες να εξισώσουν τις διαφορές, κάνετε το αντίθετο. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την, την πρωινή μας ημερήσια διάταξη και διακόπτουμε μέχρι τις 3 που θα έχουμε επανάληψη των εργασιών. Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.